Ευρώπης Λατινικής Αμερικής, ο κύριος Ταντέους Τσιμάνσκι δεν είναι πλέον τακτικό μέλος. Επίσης, έχω λάβει από το Συμβούλιο τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση μαζί με το σκεπτικό που το οδήγησε στην έγκρισή της, καθώς και τη θέση της Επιτροπής. Ο τίτλος θα ανακοινωθεί στα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης η προθεσμία των τριών μηνών την οποία διαθέτει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο προκειμένου να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο 3 Φεβρουαρίου του 2012. Θέση του Συμβουλίου εν ώψη της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών υπαριθμών 1290 του 2005 και υπαριθμών 1234 του 2007 του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Και πρώτα